ανακοίνωση στην έναρξη της ε, Τετάρτης ε, της Συνόδου του Φεβρουαρίου έλαβα αιτήματα από τους Πράσινους και από την ΓΚΟΕ